δεν προεδρεύω εγώ, αλλά είμαι εδώ για την ε, ηχογράφηση ενός ε, προγράμματος για την Ισπανική τηλεόραση και επειδή ο προεδρεύων ε, έχει καθυστερήσει για λίγα λεπτά, για να μην καθυστερήσουμε και εμείς καθυστερήσουμε και τον Επίτροπο Κάλλας, είμαι εθελοντής και αυθόρμητα για να μην καθυστερήσει η συζήτηση θα ασκήσω τα δικαιώματα του Προεδρεύοντος. Να έρθει ο κύριος Κάρας. Βλέπω ότι ένας συνάδελφος ζητά το λόγο. Και, και, no. Θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ζητήσω το λόγο στα πλαίσια του Catch αργότερα. Σήμερα το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι